7 Απριλίου στην Εστονία διορίστηκε Υπουργός Γεωργίας. Ο κύριος Αρλέμ Ντεζίρ διορίστηκε την 9η ε, Απριλίου 2014 ως ε, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η Μαρία Νταγκράσα Καρβάλιου <clears throat> θα αναλάβει το αξίωμά της ε, που με το αξίωμα του Ευρωβουλευτή δεν είναι σύμβατο. Συγχαίρω τους κυρίους Παντάρ και Ντεζίρ για τους διορισμούς τους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού